συνεδρίαση αύριο 3η 28 Απριλίου θα γίνει 8.30 με 2.30 και 3 με 11. Δημοσιεύτηκε η ημερήσια διάταξη. Είναι στη διάθεση.